ερχόμαστε στις ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε πρώτα την ε, πρόταση μορφής που κατατέθηκε κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ψηφοφορία αυτή θα γίνει με ονομαστική κλίση και χρειάζεται ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων των ε, ψηφισάντων. Παρακαλώ, καθίστε για να ψηφίσουμε. Και προετοιμαστείτε για την ονομαστική κλίση. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Μια στιγμή. Ορίστε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Σύμφωνα με τον κανονισμό απαγορεύεται να έχουμε συνθήματα πανώ ε, και τέτοια στο Κοινοβούλιο. Παρακαλώ μπορείτε να ζητήσετε ε, από τους συναδέλφους να κατεβάσουν αυτά που επιδεικνύουν. Ναι και σημαίες απαγορεύονται ξέρετε βάσει του κανονισμού. Μήπως να μαζέψετε τα σημαίακια σας. So. Λοιπόν, πέραση τη ψηφοφορία. Υπέρ 101, κατά 461, 88 εποχές. Απορρίπτεται η ε, πρόταση μορφής. So.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 Έχω και ανακοίνωση. Η διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση τη 27 Νοεμβρίου του 2014 βάσει του άρθρου 42 ε, και 45 του κανονισμού ε, και με βάση και όσα συζήτησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προχώρησε στο ε, διορισμό του κ. Τζοβάνι Μπουταρέλη